Ε, υποψήφια Επίτροπε, έτσι ολοκληρώνω το γύρο των ερωτήσεων. Μιλήσατε και μας δώσατε υπερπλήρες απαντήσεις. Αν επιθυμείτε, έχετε πέντε λεπτά για να απαντήσετε σε οτιδήποτε δεν προλάβατε να απαντήσετε και να κάνετε τα καλεκτικά σας ε, σχόλια. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά έχετε μέχρι πέντε λεπτά αν το επιθυμείτε. Επειδή πιστεύω ότι υπάρχει σε όλους μας μια κούραση, μια κόπωση μετά από τρεις ώρες, νομίζω είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο και ανθρώπινο. Θα κλείσω με δύο κουβέντες ανθρώπινες. Γιατί νομίζω αυτά που είπαμε ήταν όλα και ειλικρινή και ανταλλάξαμε καθαρές κουβέντες. Αυτή είναι, εάν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σα θα πρέπει να είναι η βάση της συνεργασίας μας. Να μιλούμε ανοιχτά, σαν μια οικογένεια. Διότι αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εσείς και εγώ είναι πολύ μεγάλες προκλήσεις. Είπε πριν ο καθηγητής δεν θα ευχόταν να ήταν στη θέση μου. Αλλά αφού μπήκαμε στην πολιτική με το πάθος της πολιτικής για να προσφέρουμε είμαστε αναγκασμένοι να μείνουμε να προσφέρουμε. Θα πω όμως κάτι που έχει σχέση με το Κοινοβούλιο γιατί νιώθω κοινοβουλευτικός. Ξεκίνησε μια διαδικασία με τις εκλογές του Μαΐου η οποία καταξίωσε την όλη εκλογική διαδικασία σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε σχέση και με τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό το hearing σήμερα ήταν μέρος αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας. Και παρόλη την κόπωση που σας είπα πριν, εν το χάρηκα γιατί ήταν ακριβώς μια δημοκρατική διαδικασία. Ήταν μια διαδικασία που καταξιώνει την πολιτική και στέλνει το μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες, εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή, τα ευρωπαϊκά όργανα, δεν χαϊδεύουμε τα αυτιά ο ένας του άλλου. Δεν στέλνουμε μεταξύ μας απλώς φιλοφρονήσεις. Κάνουμε πολιτική συζήτηση. Έχουμε πολιτικό διάλογο. Έχουμε διαφωνίες. Είπα μια διαφωνία που είχα με έναν συνάδελφο. Αλλά προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Και είναι αυτό νομίζω το βασικό επίτευγμα όλης της διαδικασίας που ξεκίνησε από τον Μάιο και θα πρέπει να συνεχιστεί. Αυτό θέλει ο Ευρωπαίος πολίτης για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του απέναντι στην Ευρώπη. Και έχουμε και οφείλουμε να του το δώσουμε. Τελειώνω με το να πω απλώς ότι πήρα πολλά σήμερα από τη συζήτηση. Έχω πολλά ακόμα να μάθω. Πάρα πολλά να μάθω. Είχα μια πολύ καλή ενημέρωση από τους ανθρώπους της Γενικής Διεύθυνσης. Τον κύριο Σόρεσεν και την ομάδα του. Τον ευχαριστώ πολύ. Δεκαπέντε μέρες δεν κοιμηθήκαμε αλλά μάθαμε κάποια πράγματα γενικά. Τώρα είναι η ώρα να μπούμε στα εξειδικευμένα, στα πιο λεπτομεριακά. Λοιπόν, νομίζω ότι εάν μου δώσετε την έγκρισή σας, μαζί θα πορευτούμε και να μάθουμε περισσότερα όλοι μας, αλλά κυρίως να κάνουμε πράξη τις απόψεις μας και το έργο μας και να κρατήσουμε την Ευρώπη ως το βασικό χορηγό ανθρωπιστικής βοήθειας για να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε Ευρωπαίοι. Thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Στυλιανίδη για την ε, τελική σας, για τα καταληκτικά σας σχόλια. Χρειάζεστε ε, ξεκούραση και την αξίζετε. Οι συντονιστές θα συνέλθουν εδώ και κλεισμένων των θύρων, γι' αυτό θα ήθελα οι μη ενδιαφερόμενοι να αποχωρήσουν από την αίθουσα. Μετά από την αποτίμησή μας θα αποστείλουμε μία επιστολή στη διάσκεψη των Προέδρων. Η διάσκεψη των Προέδρων θα κλείσει τη διαδικασία ακροάσεων. Σας ευχαριστώ όλους που προσήλθατε, ευχαριστώ και τους διερμηνείς, ευχαριστούμε και εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας, γιατί υπερβήκαμε το χρόνο, το χρόνο μας. Καλό σας βράδυ.